Καλημέρα αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καθίστε λέω και πάλι. Αρχίσαμε στις 9 το πρωί την κοινή συνεδρίαση σε άλλη αίθουσα βέβαια των ε, Επιτροπών ε, Δημοσίων Ελευθεριών και Τη Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για να συζητήσουμε το νομοθέτημα και να το ψηφίσουμε με εισηγητέ Γκρέσλε από την Επιτροπή Κοντ και εμένα προσωπικά από την Επιτροπή Λίμπερ. Τώρα επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών εδώ στην παρούσα αίθουσα. Άρα λοιπόν σας παρακαλώ Προσοχή. Συγκεντρώστε την προσοχή σας στην ημερήσια διάταξη που έχουμε σήμερα και μετά από το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ακολουθούν ψηφοφορίες. Όσοι λοιπόν εξημών έχετε τυχόν να πάρετε τις κάρτες σας, τις ηλεκτρονικές κάρτες, στείλτε κάποιον να την φέρει. Και σε αυτούς περιλαμβάνω και τον εαυτό μου βέβαια που, τις, ε, τι τις κάρτες. Ας έλθουμε λοιπόν στην ατζέντα, στην μερίσια διάταξη και πρώτα πρώτα στην έγκρισή της. Έχουν ζητηθεί κάποιες αλλαγές. Έκθεση Γκάλ για την ΣΕΠΟΛ θα γίνει θα έρθει ως πρώτη ψηφοφορία μετά το 4. Μετά έκθεση Ιντφέλτ για την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Μετά διεθνείς συμφωνίες για την ΆΣΟ. Τώρα που έχει αναβληθεί για την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Και θα γίνει και συζήτηση για την αντιπροσωπεία στη Βουλγαρία με γραπτές απαντήσεις και τον κύριο Στόγιανοφ. Και το 18 θα επιβεβαιωθεί εκεί η ψηφοφορία. Μελλοντικό γραφεία της αστυνομίας, αλλά με ερωτηματικό μετάφραση. Για το 15 στην λίστα ψηφοφορίας, λέει ο κύριος Ζάλστρα, δεν έχω λίστα ψηφοφορίας για το 15. Πότε, πότε διαβιβάστηκε αυτή. Θυμήστε μου πάλι για ποιο πράγμα μιλάτε. Α, για το Πέρικλες, για το πρόγραμμα Περικλής. Έχει διανεμηθεί θα ψηφιστεί. Εγώ δεν έχω λάβει όμως λίστα ψηφοφορίας. Δεν έχω λάβει λίστα ψηφοφορίας. Θα σας δοθεί. Θα σας δώσει η γραμματεία. Ναι κύριε Κλάις. Παρακαλώ. Ησυχία. Κύριε Μιλούμε για την ημερήσια διάταξη τώρα ή μιλούμε, ή είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Ε, ε, έθεσε ο συνάδελφό σα ερώτηση για το αν ο Περικλής θα περιληφθεί στην ψηφοφορία. Είναι λοιπόν στην λίστα ψηφοφοριών και από ό,τι μου λένε, από μου λένε διανεμήθηκε χθε με το ηλεκτρικό ταχυδρομείο. Όμω η ερώτησή μου αναφέρεται στι ανακοινώσει του Προέδρου, λέει ο κ. Κλέη. Μπορώ να την υποβάλω τώρα. Ερώτηση, ναι, ορίστε. Πρόκειται για τις ε, αποστολές αντιπροσωπιών που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες και θα γίνουν και άλλες τις επόμενες εβδομάδες. Ξαναλέω, ξαναλέω, τις τελευταίες εβδομάδες συζητήσαμε την σύνθεση αντιπροσωπιών, αντιπροσωπιών που θα μεταβούν στην Ιταλία και Βουλγαρία. Διαπιστώσαμε εμείς ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αντιπροσωπεία στην Ιταλία στη βάση του συστήματος Hunt, το οποίο εφαρμόζεται παγίως. Τώρα ξαφνικά όμως κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν εφαρμόζεται το σύστημα Hunt και θα ξαναρχίσει να εφαρμόζεται αργότερα. Γιατί δεν συνεχίζει η εφαρμογή του συστήματος Τόντ γιατί αυτή η διακοπή σημαίνει διακριτική μεταχείριση σε βάρος των μη εγγεγραμμένων. Ενώ οι μη εγγεγραμμένοι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία για την Ιταλία. Ερώτηση λοιπόν, γιατί δεν εφαρμόζονται οι κανόνες όσο εφαρμόζονταν μέχρι τώρα και όπως εφαρμόζονται και σε άλλες επιτροπές. Προφανώς κάποιοι δεν εφαρμόζουν τον κανόνα αυτόν πλέον. Και για παράδειγμα, για την αντιπροσωπεία στη Βουλγαρία, ο κύριο Σούλτς, πρόεδρος του Κοινοβουλίου, έγραψε σε επιστολή ότι ήταν υπερβολικά μεγάλη η συμμετοχή βουλευτών και αυτοί θα πρέπει να ε, πληρώσουν το ταξίδι από τα δικά τους. Κοιτάξτε, μια στιγμή, με συγχωρείτε. Κατανοήσαμε την επιχειρηματολογία σας, αλλά έχουμε ψηφοφορία. Ορισμένα μέλη έχουν έρθει μονάχα για να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Σας θυμίζω ότι την απόφαση αυτή την έλαβαν οι συντονιστές. Μπορείτε να διαφωνήσετε, αλλά οι συντονιστές αποφάσισαν ότι το σύστημα των θα γίνεται σε βάση ετήσια. Εντάξει, εντάξει. Σημειώνω, σημειώνω την άποψή σας. Επιτρέψτε, επιτρέψτε μου να συνεχίσουμε. Για το γλωσσικό καθεστώς της ε, συνεδριάσεως δεν θα υπάρξουν ορισμένες γλώσσες. Φιλανδικά, Μαλτέζικα, Κροατικά κλπ. Ο κύριος Ιακολίνο πρώτος έχει να παρουσιάσει το που βρίσκεται το θέμα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ολοκληρώσαμε άλλο τριμερή διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο κινείται τώρα προς την κατεύθυνση του κλεισίματος του σημαντικού αυτού θέματος σχετικά με την είσοδο ειδικευμένων εργαζομένων και σε ό,τι αφορά ορισμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, πολιτικών ελευθεριών, έχουμε συζητήσει και για τις ποσοστώσεις. Το κείμενο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα προνόμια και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχολήσεως, εκεί υπάρχουν ορισμένε δυσκολίες ακόμη. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ενδεδειγμένες λύσεις. στη βάση και διμερών συμφωνιών. Μιλούμε για εργαζομένους που έχουν ειδικότητε, με για παράδειγμα μάνατζερ, επίσης ε, εκπαιδευομένους σε επιπτυχίο και ούτω καθεξής, που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους εργαζόμενους υπηκόους των χωρών στις οποίες θα έλθουν να εργαστούν. διότι νομίζω ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες αποτελούν σημαντική πηγή ικανοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για την νόμιμη μετανάστευση και βάζουμε τώρα τις τελευταίες πινελιές στην, ε, ε, στο κείμενο και θα το συζητήσουν ξανά οι μόνιμοι αντιπρόσωποι. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σύντομη η παρουσίαση λοιπόν της κατάστασης μετά την, τον πρωινό τριμερή διάλογο. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία γιατί πιο πολλοί έχουν έρθει ακριβώς γι' αυτό. Έχουμε βέβαια και άλλες ψηφοφορίες. Να μην καθυστερήσουμε σχετικά σχετικά με το ΣΕΠΟΛ, είπα καταρχά στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, συνάδελφο η κυρία Κίνγκα Γκάλ, η νησηγήτρια Ξεκινάμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Πρώτο θέμα αυτό λοιπόν. Ξεκινάμε. Τροπολογία 8, απόρριψη της πρόταση, δηλαδή, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στροπολογίε, συμβιβαστική, όχι, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει συμβαστική τρία αλλά είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Κυρία Ζίπελ, τι θέλετε. Ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Ε, επειδή το συζητήσαμε ήδη αυτή την εβδομάδα ότι θα πρέπει να ζητηθεί στο μέλλον να είναι δυνατόν να γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες στην Επιτροπή. Πώς και κάνουμε τώρα ονομαστική ψηφοφορία εδώ, από όσο ξέρω δεν προβλέπεται στον κανονισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί μάλλον θα αλλάξει ο κανονισμός 50 μέλη θα μπορούν να ζητούν ονομαστική ψηφοφορία. Εδώ ζητήθηκε θα ε, γίνει η τμηματική ψηφοφορία ονομαστικά για τη συμβιβαστική τρία συγκεκριμένα. Λοιπόν, πρώτο τμήμα, ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. One PP too many. Από το ΕΛΚ ε, περισσεύουν δύο. Να βγάλουν ε, τις κάρτες τους λοιπόν από το ΕΛΚ οι παραπάνω βουλευτές. Άρχεται και περατούται ψηφοφορία. 34 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, τρίτο τμήμα έρχεται η ψηφοφορία. 32 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Μάλιστα. Πού πηγαίνουμε τώρα. Έχουν καταπέσει κάποιες τροπολογίες και περνάμε στην τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελογικέ σκέψεις τώρα. Συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική μη υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Την Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23, α όχι, συγγνώμη. Τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 23. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Καταπίπτει. Το ξεχνάμε. Πηγαίνουμε λοιπόν στην τροπολογία 4. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Όχι, όχι, όχι, καταπίπτει και αυτό. Έξι τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η επτά καταπίπτει, άρα πηγαίνουμε στο κείμενο τώρα όπως τροποποιήθηκε και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 14 κατά μια αποχή εγκρίνεται. Η εντολή τώρα για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Χρειάζεται για αυτό η ειδική πλειοψηφία. Με 31 απορρίπτεται, ψήφους αλλιώ όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Το πετύχαμε 36 ψήφοι υπέρ, 10 κατά 3 αποχές. Καλημέρα. Γεια σου. μπορώ να ξεκινήσω, λοιπόν οι διαπραγματεύσεις. Παρακαλώ, ναι, κυρία Γκάλ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στους Κιώδης και στη Γραμματεία. Πάρα πολύ επαγγελματικά εργάστηκαν όλοι για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Please let me announce the following vote, which is... Δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα, Σόφι Ιντφελντ είναι η συγγήτρια. Η τροπολογία 72 έχει αποσυρθεί. Δεν θα τη θέσω σε ψηφοφορία επομένως. Περνάμε στην τροπολογία 37 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίντ. Α, όχι, θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν 37 τροπολογία έρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Closed. Πέρας ψηφοφορίας, 28 ψήφοι υπέρ 19 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 38 ψήφοι υπέρ. 38. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε λέγω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία στα γερμανικά ο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 κατά αποχές εγκρίνεται, 61 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 64 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έχει αποσυρθεί, είπαμε. 73 και 74. Από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ, ελέγχουμε, ελέγχουμε την 81. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Λυπούμε. 82 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχής. εγκρίνεται 84. Ναι, ναι, ναι, να ελέγξουμε, να ελέγξουμε και πάλι. Την 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 23 κατά 3 αποχές. Ορίστε. 84 έτσι τώρα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Όχι, εντάξει, να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται 24 όλα. <coughs> Πάλι Μία ψήφο μα τα χάλεσε εδώ, μα την πέρδεψε. Λοιπόν, για να ψηφίσουμε τολικές αναφορέ και σκέψει. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ. να ελέγξουμε πριν ξαναγίνει τίποτα. Πριν μου φωνάξετε Εσεί, σα το λέω από μόνο. μου. Ελέγχουμε λοιπόν, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 29 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Ε, Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχή. Τι κάνετε εσείς από τη σοσιαλιστική ομάδα, να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. Είμαστε πού, Εγκρίνεται είπαμε. Δεν είναι σαφές, λέει η κυρία Ιντβέλτ. Τι ψηφίζουμε δεν, δεν έχουμε καταλάβει. Πρόεδρος, την τροπολογία 4. Λοιπόν, να επαναλάβω ή να ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε λοιπόν απευθείας την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά δεν σηκώθηκε κανένα. Ε, δεν σηκώθηκε κανένα το χέρι του από του σοσιαλιστέ και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Αλλά λοιπόν, Κλείνει η ψηφοφορία για να δούμε τι έχουμε. Πράγματι εγκρίνεται. 36 ψήφοι υπέρ 13, κατά. Τώρα το πλοίο 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίε 9 και 10. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Όχι. Να ελέγξουμε. Τις δύο αυτές τροπολογίες 9 και 10. 9 και 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ 25 κατά εγκρίνονται. Καταπίπτει 11. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 12. Πέρασε. Πέρασε είπα. 27 υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές ούτε αυτή τη φορά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Όχι. Δεν σας τα είπα καλά. Τέλος πάντων 18 υπέρ 33 κατά, αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας, γιατί εντάξει κουράζεστε, αλλά δεν είναι σαφή ε, τα αποτελέσματα μετά. Λοιπόν, τροπολογία 14, η 13 απορρίφθηκε. 14 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Όχι, ελέγχουμε, ελέγχουμε τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 23 υπέρ, 28 κατά. Λοιπόν, τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε τη 15. Ελέγχουμε τη 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 21 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Έχει ψηφιστεί ήδη. Το ίδιο ισχύει με την 18. Άρα, τροπολογία 19. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 έχει ψηφιστεί, 22 το ίδιο, 23 το ίδιο, 24 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 30 Α, όχι, 29, συγγνώμη, δεν έχει καταπέσει. 29. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 31. ΠΕΡ. Κατά αποχές απορρίπτεται 32. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 33. 33 υπέρ όχι, να ελέγξουμε την 32, το άκουσα, συγγνώμη. Ελέγχουμε. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ...29 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 34 υπέρ, Θέλετε να ελέγξουμε την 33. Ελέγχουμε. Αυτό δεν είπατε. 33 λοιπόν ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. «24 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται». Επομένως, περνάμε στην 34 ψήφι υπέρ. αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Δεν την ψηφίσαμε. Την ψηφίσαμε. Καταπίπτει, δεν καταλαβαίνω. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε, κύριος Μισελ. Για κάποιο λόγο κάποιοι πέντε συγκεκριμένα άνθρωποι δεν ψηφίζουν. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πιέστε το κομβίο παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ 18 κατά 7 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Thank you. Now, thank you, Mrs. Ευχαριστώ και την κυρία Ιντβέλτ. Θα περάσουμε τώρα στην πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Γιακολίνο είναι ο εισηγητής. Υπάρχει μια διόρθωση στον κατάλογο ψηφοφορία <clears throat> Στο 11, συμβιβαστική 11 καλύπτεται από τη συμβιβαστική 8. 27 πρώτη ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Φτάνουμε στην 33 υπέρ. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 33 ψηφίζεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας είχε απορριφθεί. Ψηφίζουμε τώρα την 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51. Κατά. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 25 υπέρ 20 κατά γίνεται δεκτή. Η Γιούρι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τζούρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή Δε, α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 86 ψηφίζεται Now closed. Πέραση της ψηφοφορίας. 21 υπέρ 24 κατά απερίφθη. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 90 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονικός έλεγχος για την 90 ψηφίζεται. Τέλος. Ξεκάθαρο, 40 υπέρ, 5 κατά, αλλά να σηκώνετε τα χέρια σας. Περνάμε στην 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 92. Ψηφίζετε. Απερίφθη. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Λοιπόν, κοντ 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 105 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 105 ψηφίζεται. Απορρίπτεται έτσι κι αλλιώς. πέρα της ψηφοφορίας. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίζει ποιος. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ δεκτή. Budget 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την budget 2. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 23 υπέρ 21 κατά. Budget 3 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι. Budget 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Γιούρι 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Γιούρι 5 υπέρ κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη Γιούρι 5 e ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Budget 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος για το budget 6. Ψηφίζεται. Τέλος. «25 υπέρ 18 κατά δεκτή». «Κοντ 2». Υπάρχει μια καταδιέρεση ψηφοφορία εδώ. ή μάλλον μόνο το δεύτερο ε, τμήμα θα ψηφιστεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κοντ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πάντζεντε 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάντζετ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την Γιούρι 7 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Γιούρι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Γιούρι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη Γιούρι 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τις ψηφοφορίες. απορρίπτεται. Κοντ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την κοντ 5 ψηφίζεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Κοντ 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της Κοντ 6. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ή δεκτή. Κοντ 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοντ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 111 είπε, κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 111 ψηφίζεται 23 υπέρ 20 κατά. Δεκτή. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κοντ 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της ΚΟΝΤ 16. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Κόντ 17 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την κοντ 17. Τέλος. 21 υπέρ, 20 κατά. Δεκτή. Α, συμβιβαστική 17 τώρα. Συμβιβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Λοιπόν, 116-125 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 17 ψηφίζεται. Ο κύριος Άλμπρεχτ θέλει το λόγο. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η γραμματεία, αλλά το δικαίωμα να ζητείτε έλεγχος ανήκει αποκλειστικά στους βουλευτές και μόνον σε αυτούς. I mean, I, I, every, every single time I've heard check, Κάθε φορά που μου λένε τσεκ λέει ο πρόεδρος, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ένας βουλευτής το ζητά. Όταν ακούω τσεκ, εν πάση περιπτώσει εννοώ ότι ένας βουλευτής το έχει ζητήσει. Εν πάση περιπτώσει έλεγχος ψηφίζουμε. Τέλο is Τέλος της ψηφοφορίας. <laughs> Well, we're, 17, no? we're, talking, we're talking 17, 17 Brigitte Sippel's amendment. Την 17 τη Sippel. Τέλος της ψηφοφορίας για την 17. Απερίφθη. Περνάμε στην 19, υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 19. Ψηφίζουμε. open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. «27 υπέρ 13 κατά, η 19 γίνεται δεκτή». Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν καταλαβαίνω τι ψηφίζετε. Εκτός αν ελέγχουμε συνεχώς ηλεκτρονικά, μήπως είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, αιτιολογική α υπέρ κατά απορρίπτεται. Β υπέρ κατά δεκτή γάμα υπέρ κατά αποχές δεκτή αιτιολογία αλφα γιούρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 25 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Το τροποποιημένο κείμενο ψηφίζουμε. πέρα ψηφοφορίας. 34 υπέρ 7 κατά μία αποχή συγχαρητήρια κύριε Γιακολίνο. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία τώρα για τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών. Το κείμενο στο οποίο, για το οποίο διαπραγματεύθηκαν στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου έλεγχος Για μια στιγμή λέει η γραμματεία, σταματάει την ψηφοφορία ο πρόεδρος. Λείπουν κάποιες ψήφοι. Μήπως κανείς αποχώρησε από την αίθουσα, φαίνεται να λείπουν τρεις ψήφοι. Τώρα όμως λίγη ψηφοφορία, λήξεις. 35 υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές. Εγκρίνεται και ευχαριστώ τον κύριο Κοέγιο για το θέμα της εποπτείας. Κυρία Μαρία Γκαμπριέλ, δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες για το σχέδιο συστάσεως. Μία ψηφοφορία μόνο, αρχίζει τώρα. Α, δύο λέτε, μάλιστα, μια στιγμή. Υπάρχει το σχέδιο συστάσεως. Εδώ αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι, ακούγεται από κάτω. Μιλούμε για την εκθεσή για την επανεισδοχή στο Αζερβαϊτζάν. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν. Λήξη. 30 ψήφοι υπέρ και 7 κατά και μια αποχή. Εγκρίνεται τώρα. Η δεύτερη έκθεση Μαρία Γκαμπριέλ. Σχέδιο συστάσεως για την διευκόλυνση εκδόσεως προξενικών θεωρήσεων. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Λήξη. 32 υπέρ 4 κατά και μια αποχή. Ευχαριστώ την κυρία Γκαβριέλ. Καλά, έγινε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε το κείμενο. Τώρα, ας δούμε άλλη ψηφοφορία με ναι. συγήτρια την κυρία Αυστέντια Σιμιέρα για κανονισμό, για ανταλλαγή ε, πληροφοριών κλπ. για την προστασία του ευρώ από παραχαράξεις. Ψηφίζουμε το κείμενο ως έχει. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Λήξη. ...38 υπέρ, 0 αποχές και 0 ψήφι κατά. Τέτοια ομοφωνία. Άρα η Τάνια Φαγιών για την διέλευση εξωτερικών συνόρων για πρόσωπα που έρχονται από χώρες που εξαιρούνται τις υποχρέωσεις έκδοσης προξενικής θεωρήσεως. Ψηφίζουμε το κείμενο που προέκυψε από τον τριμερή διάλογο. Και τώρα ψηφίζουμε. Αρχίζει. Λήξη. Ψήφι 33 υπέρ, τέσσερις κατά και μια αποχή. Και τώρα έκθεση McIntyre για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων με ποινικά μέσα για το αποτέλεσμα του ημερούς διαλόγου. Αρχίζει πάλι η ψηφοφορία. Λήξη. 37 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Ευχαριστώ την κυρία Μακιντάρ. Μία ακόμα ψηφοφορία παραμένει. Πρόταση ψηφίσματος. Α, όχι ψηφοφορία. Ναι, μα είναι ψηφοφορία. Μα το έχω και στην λίστα μου. Ας ψηφίσουμε λοιπόν το κείμενο όπως είναι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη. Το αποτέλεσμα είναι 32 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Αυτά λοιπόν για τις ψηφοφορίες. Ας συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. το υπαριθμόν 19. Όσοι αποχωρείτε από την αίθουσα παρακαλώ να το πράξετε ησύχω. Παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. the Παρακαλούνται και πάλι όσοι αποχωρούν να το πράξουν ησύχως για να προλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι που μένουμε την υπόλοιπη μερίσια διάταξη. Okay. There we go. Καλά λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Το υπαριθμόν 19. Διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 έως 20. Διδάγματα που πρέπει να αντιληθούν και οι μελλοντικέ προοπτικές. Με εισηγήτρια την κυρία Κίνγκα Γκόνς που θα εξηγήσει τη στάση τηρή για τις τροπολογίες. Αυτά λοιπόν ας... Α, μια στιγμή λέει πρόεδρο, σας παρακαλώ. Προσέξτε. Η κυρία Γκένς έχει το λόγο. Έχει το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη θα είμαι. Συντάξαμε γνωμοδότηση στην βάση των εισρώων από τους διάφορους ε, διαπραγματευτές για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά από τη συλλογή αυτή των ε, απόψεων δεν έχουμε λάβει πολλές, υπερβολικά πολλές τροπολογίες, 13 είναι όλες, και όλες. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι και επίμαχες και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Ίσως να μπορέσουμε να καταλήξουμε μάλιστα σε μία συμβαστική τροπολογία. Υπάρχει μία τροπολογία που ίσως προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων ε, πολιτικών ομάδων. Η γνωμοδότηση της Λαμπέρ, η Λάμπερτ, για το ζήτημα του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης που λέμε να μην χρησιμοποιηθεί οι πορισμένες συνθήκες και για εξωτερικές δράσεις. Εσείς δεν προτείνετε ή λέτε εκφράζει τη λύπη του που η Κομισιόν και το Συμβούλιο ζήτησαν την χρήση του Ταμείου αυτού για την χρηματοδότηση δράσεων σε τρίτες χώρες διότι αυτό αφήνει το Κοινοβούλιο χωρίς τη δυνατότητα να αντιταχθεί, να προσφύγει κατά της ε, προθέσεως αυτής. Αυτό είναι όλο που ε, συζητούμε, αν δηλαδή θα χρηματοδοτούνται εξωτερικές δράσεις ή όχι. Είναι το μόνο ερώτημα που μένει ακόμη εκρεμές. Για, τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες τροπολογίες μπορούμε να τις ψηφίσουμε την επομένη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ κυρία Γκένς για την εξήγηση των, των ε, τροπολογιών. Κυρία Τζιν Λάμπερτ. Νομίζω ναι πρέπει να λάβω το λόγο κύριε Πρόεδρε διότι η υπαριθμόν 5 την οποία μόλις ανέφερε η κυρία Γκόνς για μας εκεί το πιο σημαντικό δεν είναι απαραίτητα το περιεχόμενο Τη ουσία δηλαδή, αλλά επειδή Κομισιόν και Συμβούλιο έχουν κάνει την πρόταση αυτή, θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο μένει πλέον χωρίς κανένα μέσον να προσφύγει κατά. Όπως λοιπόν τα χειρίστηκαν τα πράγματα, λήφθηκαν ορισμένε αποφάσεις και για άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου το Κοινοβούλιο δεν μπορεί πλέον να προσφύγει κατά τις αποφάσεις του Συμβουλίου ή να αντιταχθεί τέλο πάντων. Και αυτό ανησυχεί ορισμένε και ορισμένου από εμά. Όταν θα εξετάσετε λοιπόν τις τροπολογίες μας, κοιτάξτε καλύτερα το τελευταίο μέρος της τροπολογίας παριθμών 5 και όχι την ουσία. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μελίντα Τάικ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να σχολιάσω σύντομα. Να πω πρώτα ότι μας ικανοποιεί η ιδέα να διδαχθούμε, να αντλήσουμε διδάγματα από την διαδικασία του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου είναι σωστό να δούμε ποια πράγματα απέδωσαν, ποια όχι κτλ. και στα πλαίσια των προτάσεων αλλά και σε ό,τι αφορά την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τα θέματα και τα τρία θεσμικά όργανα. Με την ευκαιρία ορισμένα σχόλια. Το ψήφισμα δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο χορήγησε η Επιτροπή πληροφορίε στο Συμβούλιο και στον τρόπο τον οποίο πληροφόρησε το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι αληθές. Εμείς φροντίσαμε οι πληροφορίε για τα χρήματα να διαβιβάζονται και στα δύο θεσμικά όργανα ταυτόχρονα. Και όντας το αρμόδιο πρόσωπο στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών φρόντισα να χορηγώ τις προφορίες αυτές και στην Προεδρία του Συμβουλίου αλλά και στη Γραμματεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ταυτόχρονα για το πώς θα γίνουν οι σχετικές περικοπές. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι δική της επιλογή, αλλά πάντως εμείς φροντίσαμε οι πληροφορίε που δόθηκαν στο Συμβούλιο να δίνονται και στο Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι είναι δύσκολο για όλους να δεχθούν τις περικοπές, αλλά παρακαλώ δείξτε κατανόηση και να είστε βέβαιοι ότι και όλοι οι συνάδελφοί μου που ορισμένοι από αυτούς είναι παρόντες εδώ συναντήθηκαν και συζητήσαν και με τους ε, εισηγητές σας, όλους τους εισηγητές για να τους ενημερώσουν. Τώρα, ορισμένα πράγματα για τις τροπολογίες, αν μου επιτρέπετε. Το Κοινοβούλιο βέβαια ακόμη δεν έχει ε, κάνει την τελική ψηφοφορία για το συνολικό πακέτο Εάν το Κοινοβούλιο λοιπόν δεν είναι ικανοποιημένο, έχει ακόμη τη δυνατότητα να καταψηφίζει, να καταψηφίσει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για τις εσωτερικές υποθέσεις. Το κείμενο βέβαια έχει συζητηθεί και τώρα βρίσκεται στα χέρια των γλωσσομαθών νομικών. Τώρα, γι' αυτό που είπε η κυρία Λάμπερτ, τη σχετική τροπολογία. Στην πρότασή της του 2011 για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε για ποιο λόγο εντός κάποιων ορίων θα ήταν σωστό να χρησιμοποιούνται χρήματα του Ταμείου και εκτός των συνόρων όπου θα έχει ενδιαφέρον για τις πολιτικές εσωτερικών υποθέσεων. Θα είναι περιορισμένο και δεν θα επικαλύπτεται με τα δραστηριότητες που χρηματοδοτούν τα άλλα ταμεία τις εξωτερικές δράσεις δηλαδή. Αυτό συζητήθηκε και προχωρήσαμε μετά στον τριμερή διάλογο. Η νομική βάση είναι αυτή την οποία θα ψηφίζετε εσείς στη Σύνοδο του Μαρτίου. Το άλλο θέμα όπου διαφωνώ είναι το, η τροπολογία υπαρθμών 6, η οποία τροπολογία λέει ότι σύμφωνα με τη συνθήκη τα εθνικά προγράμματα υπό το ΠΔΠ μπορούν να εγκρίνονται με κατεξουσιοδότηση πράξη. Δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η νομική της υπηρεσία. Εγώ δεν έχω δει ακόμα καμία, νομική γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και το συζητήσαμε διαμακρόν. Το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε στην ε, τροπολογία λέει ότι η κατεξουσιοδότηση πράξη δεν μπορούν να τροποποιούν ουσιώδη στοιχεία του νομοθετήματος. Δεν νομίζουμε εμεί ότι τούτα εδώ μπορούν να πίπτουν σε αυτό. Δεν αναμένουμε οι αποφάσεις για τα μία ταμεία να εγκρίνονται με, οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, προσπαθούμε να αποφύγουμε κάποια έγκριση στην υιοθέτηση, να οδηγήσει σε έγκριση να οδηγήσει σε καθυστέρηση μάλλον της έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων, ενώ τα κονδύλια πρέπει να ρέουν ήδη από φέτος. Και στην επόμενη συνάντησή της η Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών θα ακούσει θα ακούσει από τον αρμόδιο και εμείς βέβαια τα έχουμε πει αυτά και στην Προεδρία της ε, Επιτροπής αλλά και στις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστως θα προσέρχεται τακτικά ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών σε όλη την διάρκεια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου για να σας ενημερώνουμε και να ακούμε τις ανησυχίες σας και ή δυνατόν να διαφθώσουμε ένα διάλογο για την ε, εφαρμογή των κονδυλίων και την χρήση των κονδυλίων του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Βεβαίω δικό σα είναι το ψήφισμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι δίνει κάπω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε μονόπλευρη. Έχω δίπλα μου ωστόσο το μέλο τη Ελληνική Προεδρία και μπορώ να σα βεβαιώσω ότι οποιαδήποτε χώρα μέλο η οποία συμμετέσχε στη συζητήση του Συμβουλίου δεν είχε καθόλου την εντύπωση ότι η Κομισιόν συμπαρατάχθηκε αποκλειστικά μαζί του. Και σε όλε τι διαπραγματεύσει εμεί προειδοποίησαμε το Συμβούλιο να μην λάβει αποφάσει που ενδεχομένω θα καθιστούσε δυσχερή την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε και στις υποχρεώσεις μας από τη συνθήκη και απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα με πλήρη σεβασμό προς το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Κυρία Γκέντς, να μας ξαναπεί. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπατε κι εσείς, ότι δηλαδή την, υπάρχει αυτή η έκθεση ε, της Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου. Εγώ δεν συμμετείχα στο σύνολο των διαπραγματεύσεων, αλλά σε μέρος των διαπραγματεύσεων. Και όπως είπα και στην αρχή, αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν να ρωτήσω τους συναδέλφους μου. Και το σχέδιο έκθεσης ε, ουσιαστικά αποτελεί μια αποδεκτή ε, γνωμοδότηση. Αποδεκτή από τους περισσότερους από όσους συμμετείχαν και θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών από την Κομισιόν με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό το άκουσα από πολλούς από τους ε, συναδέλφους οι οποίοι διαπραγματεύονταν ε, τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις απαντήσεις σας και για την ε, απόψή σας για το πώς βλέπετε την όλη διαδικασία. δεν ξέρω αν αληθεύει ότι έλαβαν στο Συμβούλιο περισσότερες πληροφορίες, δεν διατυπώθηκαν πάντως παράπονα. Δεν ξέρω αν υπήρχε αντίθετη εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο παίρνει περισσότερες πληροφορίες, ίσως να είχαν διαμαρτυρηθεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτό ε, το σχέδιο έκθεσης αντικατοπτρίζει τις απόψεις του Κοινοβουλίου, των συναδέλφων που συμμετείχαν, Καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά ε, το θέμα είναι να μην διαμορφώνεται μια τέτοια εντύπωση, γιατί αυτή την εντύπωση έχει διαμορφώσει το Κοινοβούλιο. Από ό,τι βλέπω, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε την έκθεση, γιατί υπάρχει ευρύτατη υποστήριξη. Έγινε μια μακροσκελέστατη συζήτηση για την ερμηνεία των κατεξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και οι διάφορες αστυνομικέ υπηρεσίε έδωσαν διαφορετικές ερμηνείες. Εκτιμούμε λοιπόν τη δική σας άποψη. Τι δεχόμαστε μένα, αλλά εμείς προχωρούμε με τη δική μας ε, έκθεση, που είναι και, όπως είπα, η άποψη των διαπραγματευτών για την ε, Jean Lambert. Είναι ευρέως αποδεκτή αυτή η άποψη, ότι η διαδικασία δεν θεωρήθηκε δίκαιη ή ισορροπημένη από αυτήν την έννοια. Αυτό άκουσα τουλάχιστον από πολλούς συναδέλφους θεωρούσαν ότι ήταν ήδη έτοιμη αυτή η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν, άρα δεν είχε λόγο ουσιαστικά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο. Το άλλο θέμα βέβαια είναι για το αν θα χρησιμοποιήσουμε για τις εξωτερικές σχέσεις. Σας ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τη Δευτέρα, Πρόεδρος είδα ε, να σηκώνει το χέρι ένας άλλος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να διευκρινίσετε κάτι. Θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας. Ευχαριστώ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνη. Θα ήθελα να πω για τα θέματα που αφορούν ε, τη δικαιοσύνη, αφού η έκθεση πραγματεύεται και τα δύο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τις ε, επικοδομητικές διαπραγματεύσεις που είχαμε. Και έτσι θα μπορέσ, μπόρεσαν να εγκριθούν και οι δύο κανονισμοί στα τέλη του 2013, γέρος δηλαδή. Και στους συνομοθέτες και τους δύο ε, διβάσαμε την έκθεσή μας. Εμείς τώρα επεξεργαζόμαστε τα ειδήσια προγράμματα να σας πω ότι θα έχουμε σύντομα προκήρυξη διαγωνισμών και θα συμπεριλάβουμε στις υποχρεώσεις μας για την ετήσια υποβολή εκθέσεων και τους μηχανισμούς ε, ε, υποβολής εκθέσεων, reporter Ναι, χαίρομαι πιστεύω γιατί υπήρχε ένα θέμα, υπήρχε μια διαφορά μεταξύ των φακέλων που αφορούν στις ιστορικές υποθέσεις και των φακέλων που αφορούν ε, τη δικαιοσύνη. Είχα πολύ θετική εμπειρία συνεργαζόμενη με την Κομισιόν. Το είπα και πριν ότι ήταν πολύ δημιουργική η προσέγγιση της Κομισιόν και μπορέσαμε να εργαστούμε πολύ καλά. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Χαίρομαι, δεν σας είχα δει νωρίτερα, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Ναι, πράγματι καλό ήταν να ακουστούν και οι δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης. Oh, Ολοκληρώνουμε λοιπόν με το θέμα αυτό προ το παρόν το επόμενο σημείο. Υποτίθεται θα συζητούσαμε στις 12 παρα 20 και θα έχει ως αντικείμενο αυτό το θέμα την αντιπροσωπεία στη Βουλγαρία ο εισηγητής επικεφαλής αντιπροσωπείας αυτής δεν είχε έρθει ακόμη γιατί περίμενε ότι θα συζητηθεί το θέμα στις 12 παρα 20, άρα κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών και θα επαναλάβουμε στη συνέχεια τις εργασίες μας.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Σεβεά και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

Ε, I would like to welcome everyone who came back after the... Να σας καλωσορίσω όλους όσοι επιστρέψατε μετά το διάλειμμα να ζητήσω από τους συναδέλφους να καθίσουν για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Αντιπροσωπεία στη Βουλγαρία και κατάσταση αυτών που ζητούν άσυλο και πρόσφυγες από τη Συρία. Έγινε η επίσκεψη στις 20 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου. μαζί με την ερώτηση του κυρίου Στογιάνοφ. Θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από τον κύριο Έγκελ ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της αντιπροσωπείας, να μας δώσει μία περίληψη. Και η κυρία Γκυγιόμ είχε πάει εκεί, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Γι' αυτό ο κύριος Τέγκερ θα μας ενημερώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι Είχα 50% πιθανότητες να είμαι υπεύθυνο της αντιπροσωπείας γιατί δύο ήμασταν. Αλλά είχαμε και πολλούς βούλγαρους συναδέλφους οι οποίοι μας συνόδευσαν. Δεν ξέρω πόσο έχει κυκλοφορήσει η έκθεση και πόσο είναι διαθέσιμη. Κανονικά πρέπει να είναι σε όλους διαθέσιμη. Είχαμε ένα πληρέστατο πρόγραμμα. και για την εξέλιξη της κατάστασης και για την εισρωή προσφύγων από τη Συρία, κυρίως από τη Συρία αλλά όχι μόνο από τη Συρία. Είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε επίσης και κάποια πιο κρίσιμα σημεία για τις υποδομές υποδοχής αυτών που έρχονται στη Βουλγαρία ζητώντας διεθνή προστασία. Αυτοί δεν θέλουν όλοι να μείνουν στη Βουλγαρία βέβαια, δεν θέλουν να έρθουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βουλγαρία επειδή βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όλος τυχαίως, είναι προφανές ότι είναι ένα από τα πρώτα εδάφη στα οποία πηγαίνουν οι υποψήφοι αυτοί πρόσφυγες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι η Βουλγαρία ε, δεν ήταν και εξακολουθεί εν μέρη να μην είναι ιδανικά προετοιμασμένη για την υποδοχή τέτοιου είδους ανθρώπων και για την παροχή προστασίας όταν υπάρχει μια μείζον κρίση όπως η Συρία και μετά από όλες τις άλλες αναστατώσεις στην περιοχή, έχει κανείς να αντιμετωπίσει με τόσο μεγάλους αριθμούς που αμφιβάλλω αν η αδίποτε άλλη χώρα θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει κάτω από καλύτερες συνθήκες. Βελτιώνονται τα πράγματα πάντως. Πιστήκαμε γι' αυτό ότι λαμβάνονται περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση των μέτρων υποδοχής, θα πρέπει να περιμένουμε. Και στην περίπτωση που υπάρξουν στο μέλλον δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον προσφύγων, που περάσουν τα βουλγαρικά σύνορα, προφανώς το θέμα των συνθήκων υποδοχής και των υποδομών υποδοχής ε, θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβληματισμό. Αυτά για τους αριθμούς που ε, ε, αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εγκαταστάσεις υποδοχής που μπορεί να υποδεχθούν το πολύ 35.000 κόσμου όλων των κατηγοριών. Γνωρίζουμε ότι στην Τουρκία μόνο υπάρχουν γύρω στους 750.000 Σύρους. Και άλλοι τόσοι στο Λίβανο. Και φυσικά υπάρχουν και εκατομμύρια Σύροι εκτοπισμένοι στο εξωτερικό της χώρας που θα ήθελα να πάνε αλλού για να ξεκινήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Και γι' αυτό είπαμε και στο πρώτο σημείο των συμπερασμάτων ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζει. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τη Βουλγαρία όταν οι συνθήκες υποδοχής ε, δεν είναι καλές. Όταν δεν γνωρίζουμε πόσους σύρους θα ήθελε να καλωσορίσει η υπόλοιπη Ευρώπη στην περίπτωση που αυξηθούν οι αριθμοί στα επίπεδα τα οποία αναφέραμε. Ακούω για λίγες εκατοντάδες. Η Γαλλία λέει θα υποδεχθεί 500. 60 η δική μου χώρα, 28 σύντομα. Αλλά αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν καμία σχέση με τους αριθμούς που μας αφορούν τώρα. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η κρίση δεν πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω και ακόμα και αν υπάρξει μια ρύθμιση στη Συρία δεν ξέρω τι θα γίνει στη Λιβύη αύριο και στις υπόλοιπες χώρες γύρω μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για να φιλοξενήσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν αποφασίζουν από μόνοι τους να φύγουν αλλά είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να πάνε κάπου αλλού γιατί η ζωή τους είναι σε κίνδυνο και δεν υπάρχει τίποτα πια για αυτούς. Και ένα πολιτισμένο περιβάλλον όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> πρέπει να προετοιμαστεί να τους υποδεχθεί, αν χρειαστεί. Δεν θέλω να παρατείνω λοιπόν την παρουσίασή μου. Εμείς προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τις συνθήκες υποδοχής δεν ήταν πολύ καλές, εξελίσσονται θετικά, υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως και σε όλες τις άλλες χώρες. Τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς όταν εγκαταλείπουν τα κέντρα υποδοχής, χάνουν το καθεστώς προστασίας που είχαν. Από ό,τι φαίνεται στην παρούσα φάση η Βουλγαρία έχει να κάνει με πάρα πολύ ε, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι αμόρφωτοι, είναι αναλφάβητοι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους ενσωματώσει κανείς ε, και στην αγορά εργασίας ε, και στην κοινωνία γενικότερα. Γι' αυτό το θέμα της ενσωμάτωσής τους τίθεται και από τις αρχές σιγά σιγά, αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα. Ένα άλλο θέμα μεγεθυνθεί είναι οι ασυνόδευτοι ε, νέοι, τα παιδιά, ανήλικοι. Δεν είδαμε, εμεί είχαμε ακούσει αριθμούς αλλά δεν είδαμε τέτοιες περιπτώσεις και από όσους ρωτήσαμε δεν είχαν και αυτή υπόψη. Υπάρχει υποτίθεται ένα ειδικό κέντρο το οποίο δεν μας προβληματίζει αφ' αυτού, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει στο μέλλον. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο δείχνει το υψηλό επίπεδο υποκρισίας το οποίο επιδεικνύει η Ευρώπη. Κατηγορούνται οι Βούλγαροι γιατί δημιουργούν ένα φράκτη στα σύνορα με την Τουρκία. Οι αρχές ισχυρίζονται διάφορα τα οποία δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε. Ότι είναι επικίνδυνα τα εδάφη αυτά και ότι στην ουσία παρέχεται μια κάποια προστασία. Κοιτάξτε, βρίσκω λογικό η Βουλγαρία να προστατεύει τα σύνορά της γιατί της το ζητάμε, της το απαιτούμε αυτό στα πλαίσια και της ένταξής της στο χώρο Σέγγεν και ταυτόχρονα καταδικάζουμε τη Βουλγαρία γιατί στερεί τη δυνατότητα σε ανθρώπους να μπουν στο έδαφος της το οποίο είναι βέβαια μια διεθνής ανηλυμένη υποχρέωση. Κάτω από δίποτες συνθήκες δεν ισχύει κάτι τέτοιο όμως είπε η Βουλγαρία ότι υπάρχουν σημεία εισόδου επίσημα, τελωνιακή σταθμή και ότι κάποιοι οι οποίοι παρουσιάζονται εκεί και μπορούν να τύχουν υποδοχής. Θυμίζω ότι ένας τέτοιος φράκτης υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα είχαμε λιγότερα προβλήματα με το φράκτη αυτό από ό,τι έχουμε τώρα με τη Βουλγαρία όπου δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις βέβαια. Μια κρίσιμη γεωγραφική θέση που κάνει τη χώρα αυτή να είναι εκτεθειμένη σε μεταναστευτικές πιέσεις πιο σημαντικές από όλες οι άλλες χώρες, οι εσωτερικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται το θέμα της ικανότητας των βουλγαρικών αρχών να ελέγχουν, να αστυνομεύουν και να διασφαλίζουν τα σύνορά τους, τα εξωτερικά, να επιτρέπουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και που ζητούν διεθνή προστασία να μπαίνουν στη Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος η αντικειμενική ανάγκη μιας ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του προβλήματος γιατί καμία χώρα και μάλιστα οι φτωχότερες της Ένωσης δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους τέτοιου είδους ε, μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουμε εκ νέου στο μέλλον και τους επόμενους μήνες. Τέλος, η Βουλγαρία έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής των προσφύγων. Δεν αρκούν, αλλά συνεχίζονται. Αυτό το παράδειγμα είναι μια επιπλέον έκκληση σαν και αυτές ε, που έγιναν για τη Λαμπεντούζα και για τις υπόλοιπες ε, νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. Ακούσαμε τα ίδια και για το φαρμακονήσι στην Ελλάδα που πνίγηκαν κάποιοι πρόσφυγες ε, όπου πνίγηκαν κάποιοι πρόσφυγες λοιπόν στο μέσο μιας καταιγίδα και όπου ακούγονται πάρα πολλά σχόλια θετικά και αρνητικά για τη στάση γενικά. Στο βορρά της Ευρώπης ε, φαίνεται ότι εμείς προτιμάμε να αφήνουμε τους νότιους να ασχολούνται με τέτοια θέματα γιατί μόνο σε αυτούς συμβαίνουν. Εμείς σαν ευρωβουλευτές θα πρέπει να καταγγέλουμε το απαράδεκτο των συνθήκων υποδοχής σε οποιαδήποτε περιοχή και να αναλάβουμε επιτέλους τις ευθύνες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνοπτική αυτή παρουσίαση. Από ό,τι κατάλαβα στην επίσκεψη αυτή ήταν ξεκάθαρο πόσο αμφιλεγόμενα μηνύματα δίνονται. Δηλαδή αφενός προστασία συνόρων ε, που είναι απαραίτητη για την ένταξη της χώρας στο Σέγγεν, από την άλλη ε, να επιτραπεί ή να μην επιτραπεί είσοδο ε, στους άσυλο στη χώρα. Και αν ναι, ε, να μην ε, τους δοθεί δυνατότητα να πάνε σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες τη Ευρώπη Είναι υποκριτική αυτή η στάση. Γι' αυτό έχουμε άλλωστε και την κρίση αυτή τη στιγμή, την κρίση στη Μεσόγειο. Όπως είπα, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό από κοινού με με την Κομισιόν γιατί ζήτησε ο κύριος Στογιάνοφ μια γραπτή απάντηση από την Κομισιόν Θέλατε να το συζητήσουμε στη ή Δεν είχατε λάβει απάντηση, τώρα την έχετε λάβει, αν κατάλαβα καλά. Θα ζητήσω από την Κομισιόν παρόλα αυτά να μας παρουσιάσει συνοπτικά την απάντησή της. Και νομίζω ότι και ο κύριος Ήρθε και ο κύριος Στογιάννου θέλουν το λόγο. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Στογιάννου που ήταν και αυτός που υπέβαλε την προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 16 Οκτωβρίου έστειλε αυτή την, προφορική ερώτηση, την, συγγνώμη, την γραπτή ερώτηση στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πρόκειται ουσιαστικά για τρεις ερωτήσεις. Απλές τις θεώρησα τις ερωτήσεις και περίμενα να μου απαντήσει πολύ γρήγορα η Κομισιόν στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας. Έλαβα στις 12 Δεκεμβρίου όμως την απάντηση τελικά. Όπως γνωρίζετε, τρεις εβδομάδες ε, θα έπρεπε να είχε διαρκέσει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με την απάντηση, εξού και θέλω να λάβω το λόγο σήμερα. Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις στην απάντηση κομψή. Στην πρώτη σελίδα τη απάντηση, όταν ρω... βρίσκεται αυτή η αντίφαση, γιατί είχα ρωτήσει κατά πόσον Γι' αυτό το ταμείο για τους πρόσφυγες έχει δώσει χρήματα η Βουλγαρία. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι δεν υπάρχει ταμείο, δεν υπάρχει κονδύλια για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης της Συρίας. Από την άλλη όμως υπάρχει μια κοινή δήλωση ε, από τα κράτη-μέλη για δύο ε, εκατομμύρια. Α, συγγνώμη, δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέτε αυτά κάποιο ταμείο, δεν τα, εντάξει, δεν είναι ένα ταμείο που έχει ε, συσταθεί ad hoc. Πώ θέλετε πείτε το, αλλά υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν κονδύλια για αυτό το σκοπό. Δεν είναι λοιπόν άμεση απάντηση. Θέλει να πει η Επιτροπή ότι δεν ε, δεν έχω καταλάβει, τι να πω. Σε αυτό το μη ταμείο τέλος πάντων ε, υποτίθεται ότι έχει δώσει 300.000 η Βουλγαρία. Πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί από το ταμείο αυτό. Απαντά η Επιτροπή, καμία, μάλλον απάντηση. Επίτροπος Γεωργίευα, στην οποία έγραψα, μου λέει, ναι υπάρχει αυτό το ταμείο και το διαχειρίζομαι εγώ ως Επίτροπος. Η Επίτροπος Μάλστρομ τώρα μου λέει δεν υπάρχει τέτοιο ταμείο. Γιατί διγλωσία τέτοια. Γιατί ο ένας ή μία Επίτροπος να έρθει σε ε, να διαψεύδει την άλλη. Έχω και άλλες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα. Γιατί ε, αργείτε, γιατί κολυσιεργείτε και γιατί επεκφεύγετε. Είναι τόσο δύσκολο να γράψετε μια σελίδα, μια απάντηση. κάπως ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα η Κομισιόν, αλλά το γεγονός ότι δεν απαντά εγκαίρως, για μένα αποδεικνύει ότι η Κομισιόν δεν αναζητεί αντικειμενικές απαντήσεις, απλά τελικά μου απαντούν ως μέλος της βουλγαρικής αντιπροσωπείας, και σαν άτομο με αρρωστημένη περιέργεια. Για αυτά τα δύο δις την εκταμείευση αυτών των κονδυλίων. Μπορείτε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, πώς δαπανήθηκαν αυτοί οι πόροι. Η Βουλγαρία είναι και από τα φτωχότερα κράτη. Οι συντάξει είναι 100 ευρώ το μήνα. Έδωσε όμως 300.000 ευρώ η Βουλγαρία. Αυτή ήταν η συνεισφορά της σε αυτό το ταμείο των 2 Άρα αυτό σημαίνει συντάξει 3.000 ε, Βούλγαρων υπηκόων. να πω και ακόμα, να θέσω και άλλα δύο ερωτήματα. Αφού ευχαριστήσω τον κύριο Έγγελ, ε, θέλω να πω ότι σίγουρα η Βουλγαρία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά τη, να αστυνομεύει, να ελέγχει τα σύνορα, αλλά δεν είναι μόνο σύνορα της Βουλγαρία, είναι και σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεσμευτήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα τα διατηρήσουμε ασφαλή τα σύνορα. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει με το εξή. Είναι σαφέ ότι οι περισσότεροι από του πρόσφυγε, δεν ξέρω πόσοι είναι, γύρω στου 12.000, α πούμε ότι είναι πρόσφυγε. Είναι πρόσφυγε μεν, αλλά αποδεικνύεται τελικά ότι πρώτον δεν είναι Σύριοι και δεύτερον δεν είναι Σύριοι και αν είναι Δεν είναι πρόσφυγε. Γνωρίζουμε τι προβλέπει η διεθνής νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η απόθυση, η επαναπρόθεση. Τι κάνεις όμως όταν έχεις στα σύνορά σου έναν παράνομο μετανάστη. Δεν πρέπει η Βουλγαρία να έχει την απαιτούμενη οργάνωση ώστε να μπορεί να στέλνει στα συνοριακούς σταθμούς αυτά τα άτομα και μετά εκείνο αποφασίζει ποιος πρέπει να επαναπροωθηθεί ως λαθρομετανάστη και ποιος ε, δικαιούται να εισέλθει στη χώρα. Μια απάντηση τώρα για το άρθρο 33 και είναι και ολοκληρώνω με αυτό, για το Δουβλίνο 2 δηλαδή. Διακόπτει ο Ξέρετε, θέλετε να ακούσετε την γνώμη τη Επιτροπή, το λέτε και εσεί, αλλά μην μακρηγορείτε λοιπόν. Ναι, κύριε Στελιάν, θέλω απλά να τα διατυπώσω σωστά για να πάρω και μια ωραία απάντηση. Λοιπόν, άρθρο 33 του Δουβλίνου 2. Είναι πρόβλημα. Κάποιοι βούλγαροι συνάδελφοι είπαν δεν μπορούμε να το επικαλυστούμε αυτό το άρθρο. Γιατί αφού πρέπει να ε, επιδεικνύεται αλληλεγγύη και να εφαρμόζονται σωστές πολιτικές. Ποια είναι λοιπόν η διαδικασία του άρθρου 33 που ξέρουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα θα ήθελα να με εξηγήσετε παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριο Ήρτσεφ και μετά η Κομισιόν απαντήσει παρακαλώ. Στα δύσκολα αυτά ερωτήματα. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την έκθεση για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, ήδη από, την, από το φθινόπωρο πέρσι ήταν δική μου ιδέα η κατάσταση στη Βουλγαρία να αναλυθεί και οι σχετικές προφορίες να συζητηθούν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών σε ευρύτερο πλαίσιο, γιατί εγώ ανέμενα κλιμάκωση του προβλήματος στην Βουλγαρία, κλιμάκωση των προβλημάτων μάλιστα, προβλημάτων που ε, προέρχονται και εκτός των συνόρων της χώρας. Η αντιπροσωπεία αυτή με τον κύριο Έγγελ υπήρξε επιτυχής. Και αυτό φαίνεται και στην έκθεση. Συναντήσαμε τις σημαντικές προσωπικότητες της εκτελεστικής εξουσίας και της, και της νομοθετικής εξουσίας και άλλους. Η έκθεση είναι λεπτομερής και εμπεριστατωμένη και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ τον κύριο Έγγελ και εκφράζω την εκτίμησή μου για τις προσπάθειές του να φανεί και υπομονητικός και αποτελεσματικός. Η έκθεση θα είναι σημαντική στις επόμενες συζητήσεις που θα γίνουν στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας, γιατί οφείλω να επενθυμίσω ότι είναι πλήρης σε λεπτομέρειες παραδείγματα και συμπεράσματα. Τρία σχόλια τώρα. Πρώτο, η νομοθεσία στην Βουλγαρία χρειάζεται βελτίωση και αυτό απηχείται στην έκθεση. Χρειάζεται αλλαγές. Ιδίω, το άρθρο 35 του ισχύοντος νόμου περί ασύλου στην Βουλγαρία. Το άρθρο αυτό και ορισμένα άλλα συναφή κύματα, κείμενα συγγνώμη, χρειάζονται αλλαγή, ιδίω για τις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για επανένωση οικογενειών. Όπως βλέπετε από την έκθεση τώρα, έχουμε 192 ασυνοδεύτους ανηλίκους και πρέπει να υπολογίσετε και τη σημαντική πρόκληση για τις βουλγαρικές αρχές εάν πρόκειται να επανενώσουν τις οικογένειες αυτές. Θα πρέπει να υπολογίζουμε καμιά εξακοσαριά ε, γονείς και στενούς συγγενείς για να επανενωθούν με τα 192 αυτά ασυνόδευτα ανήλικα ε, πρόσωπα. Ο περίφημος φράχτης στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Νομίζω ότι η έκθεση αλλά και η ανάπτυξη του θέματος του κύριο Έγγελ δίνει την πλήρη απάντηση. Δεν είναι τείχος ανάμεσα σε δυο γειτονικέ χώρες, δεν είναι πρόκληση, είναι ένας ελαφράς κατασκευής φράχτης για να αποτρέψει εκείνους που θέλουν να περάσουν από σύνορα από, δύσκολους, από δύσκολα δύσβατα σημεία και να τους προσανατολίσει στα checkpoint. Οι άνθρωποι αυτοί δεν περνούν από τα checkpoint, διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να περάσουν από άλλα σημεία όπου δεν υπάρχει εποπτεία. Τέλος, Η έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες των βουλγαρικών αρχών να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Και να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε προηγούμενα γύρω από το θέμα του φράχτη. Η έκθεση, και αυτή είναι η σύστασή μου, μπορεί να διανεμηθεί και σε μέρη άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών και κυρίως στην Επιτροπή Εξωτερικών. Επίσης μπορεί να υποβληθεί και στην νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πληροφόρηση. Όλα τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως ποια είναι η κατάσταση στη Βουλγαρία. Η κυρία Κίνγκα Γκόνς που προεδρεύει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάει τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας λάβει το λόγο για να απαντήσει τις ανησυχίες καθώς και τις ερωτήσεις των μελών. Έχει το λόγο κύριε. κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τα ερωτήματα του κύριου Στογιάννοφ. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω ότι απαντήσαμε καθυστερημένα στη γραπτή σας ερώτηση και εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτό. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά ε, την υποχρέωσή μας να απαντούμε σε ερωτήσεις ε, των Ευρωβουλευτών. Προσπαθούμε πάντοτε να τηρούμε τις προθεσμίες. τι περισσότερες φορές το επιτυγχάνουμε. Ενίοτε για τις ε, απαντήσεις χρειάζεται να συνεργαστούν περισσότερα άτομα από διαφορετικές υπηρεσίες της Κομισιόν και αυτό καθυστερεί κάπως τη διαδικασία, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Προσπαθούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες, δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση όμως αργήσαμε. Να έλθω όμως στην ουσία. Ελπίζω να μην χρειαστεί να συζητήσουμε τα ζητήματα ορολογίας, να μην ε, μακρηγορήσουμε για την ορολογία, αλλά όπως απαντάμε και στην ε, γραπτή μας απάντηση, υπάρχει ένα ειδικό ταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε για τη σειρακή κρίση. Ε, υπάρχουν δαπάνες ε, από διάφορα μέρη ε, για να βοηθηθούν ε, οι πληγέντες από τη Συριακή κρίση. Ε, από αυτό προέρχεται και το συνολικό ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι το άθροισμα ε, συνολικών, των συνολικών δαπανών από διάφορες, διάφορες γραμμές ε, και από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη που ε, παρέχουν χρηματοδότηση σε χώρες όπως είναι η Ορδανία, ο Λίβανος, η Τουρκία στις αρχές των χρόνων αυτών ή σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις που επί Συνολικά η δαπάνη που προέρχεται από τα κονδύλια του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική υποστήριξη και την αναπτυξιακή βοήθεια δηλαδή, ουσιαστικά αποσκοπεί στην ε, παροχή πρακτικής βοήθειας σε αυτούς που αντιμετωπίζουν ε, την ε, κρίση των προσφύγων που προέρχονται από τη Συρία. Το ποσό που έχει διαθέσει η Βουλγαρία δεν πέρασε μέσα από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία πρόσφερε κάποια χρήματα σε άλλες χώρες της ε, περιοχής απευθείας. Δεν μπορώ να σας πω ε, ποιο ποσοστό έχει ταπανηθεί, αλλά αυτό το ποσό ε, δεν πέρασε από τις Βρυξέλλες. Αυτά για το πρώτο. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση κατά πόσον έλαβε η Βουλγαρία κονδύλια από αυτή τη δαπάνη. Όχι. Όχι από αυτά τα κονδύλια τα οποία σας αναφέρω στην απάντησή μου και τα οποία αφορούν τη δαπάνη ε, για την περιοχή της Συρίας. Στο μεταξύ όμως, και αφού σας διαβιβάσαμε την απάντησή μας, μπορούμε τώρα να προσθέσουμε ότι σε ό,τι αφορά την παροχή στήριξη στη Βουλγαρία, Το Γραφείο Στήριξης Προσφύγων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΑΣΟ, στηρίζει πλέον τις βουλγαρικές αρχές και θα ε, συνεχίσει να το πράττει σίγουρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Επίσης έχουμε δώσει κατεπίγουσα ε, χρηματοοικονομική ενίσχυση στην Βουλγαρία στο πλαίσιο του SOLID που είναι το ταμείο μας ε, για τις εσωτερικές υποθέσεις. Συνολικά 5,6 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, 2,4 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα Σύνορα και από αυτό το ποσό νομίζω ότι έχει καταβληθεί προκαταβολικά το 80%. Είναι ήδη στη Βουλγαρία και από το Ταμείο της Επιστροφής είναι λίγο παραπάνω από 500.000 ευρώ. Να ήλθω τώρα σε κάποια πιο γενικά σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνεί με πολλά από αυτά που είπε ο κ. Σέγγελ και συμμεριζόμαστε την ανησυχία των αξιότιμων ευρωβουλευτών για την πίεση, τις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχονται, ιδίω η Βουλγαρία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Οι βουλγαρικές αρχές ε, έχουν κάνει πολλά, όταν ξέσπασε η κρίση στη Συρία και σε συνεργασία με την Κομισιόν και με το ΕΑΣΟ, με την Υπατή Αρμοστή για τους πρόσφυγες, με πολλές ΜΚΟ. Πολλές ε, λοιπόν ε, είναι οι δραστηριότητες επιτόπου για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης θεωρούμε ότι τουλάχιστον έχει επέλθει σταθεροποίηση και συγκράτηση ε, της κατάστασης. Δεν επιδεινώνεται δηλαδή προς το παρόν. Ωστόσο, είναι πολλές οι προκλήσεις, σαν αυτές που μας ε, περιέγραψε και ο κύριος Έγγελ. Δηλαδή, η κατάσταση των ετούντων άσυλων και μεταναστών στα κέντρα φιλοξενίας. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στην επεξεργασία των αιτήσεων ε, ασύλου και το πώς εντάσσονται στην κοινωνία αυτοί που έχουν πλέον λάβει αυτό καθεστώς προστασίας συζητήθηκε και το άρθρο 33 του κανονισμού Δουβλίνου. Είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας είναι σαφές ότι εφόσον ενεργοποιηθεί, δηλαδή αν υπάρξει σύσταση από την Κομισιόν δυνάμει του άρθρου 33, σε κανένα περίπτωση αυτό δεν θα πρόκειται για ε, να κατηγορηθεί, να τιμωρηθεί εντό αγωγικών η Βουλγαρία οποιοδήποτε άλλο. Απλά αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό η ε, ύπαρξη του προβλήματος, ότι έχουμε μια σοβαρή κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό, ε, αυτή η σύσταση θα εκπέμψει ένα χειρό μήνυμα που θα λέει ότι δεν είναι μόνη της η Βουλγαρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη να βοηθήσει τη χώρα αυτή για ε, να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Θα σημαίνει επίσης ότι απευθύνουμε και μια διεθνή έκκληση για αλληλεγγύη με την Βουλγαρία. Ε, τόσο ηλικία όσο και επιχειρησιακή βοήθεια. Και θέλω να τονίσω ότι ήδη έχει κινητοποιήσει η Κομισιόν ε, ε, υποστήριξη και συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Τώρα, κατά πόσον θα γίνει σύσταση δυνάμει το άρθρο 33, θα το αποφασίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπως σας είπα το εξετάζει αυτή τη στιγμή και σε έφτατο χρόνο θα λάβουμε απόφαση σε επίπεδο σώματος επιτρόπων για να δούμε κατά πόσον θα γίνει ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ για την απάντησή σας. θα κάνουμε και άλλη ψηφοφορία μαζί με την Επιτροπή Οικονομικών. Να δώσω λοιπόν πάλι το λόγο σύντομα στον κύριο Έγγελ για να συνοψίσει ορισμένα πράγματα και κάτι που ήθελα να πω εγώ επίσης η πρόταση δηλαδή να διαβιβαστεί η έκθεση στην Επιτροπή Εξωτερικών και να την ε, μοιραστούμε μαζί τους, να την υποβάλουμε δηλαδή σε αυτούς. Καλή ιδέα να το αναλάβει η γραμματεία γιατί και αυτοί μπορούν να, την, μπορεί να την χρειάζονται. Φρανκ Έγγελ, γιατί έρχονται σιγά σιγά και τα υπόλοιπα μέλη για την ψηφοφορία. Ναι βεβαίως δεν θέλω να καθυστερήσω κι εγώ περισσότερο μέχρι να καθίσουν οι συνάδελφοί μου. Θα πω εγώ πρώτον ευχαριστώ στους συναδέλφους για την συζήτηση. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που έδωσε. Για την ίδια την έκθεση δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Οι περισσότεροι που τους αφορά φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι. Θα αρκεστώ σε αυτά. Η κυρία Γκόνς, σας ευχαριστώ για την εργασία που έχετε επιτελέσει για το θέμα αυτό. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το τμήμα της συνεδριάσεως. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 24 Δευτέρου στο Στρασβούργο, όπου προβλέπεται ψηφοφορία και εκεί βεβαίως παρακαλείστε να είστε παρούσες όλες. Και... και στις 10 Μαρτίου αντί τις 6. Έχω εδώ 6 και θα έχουμε και την κοινή συνεδρίαση. Βλέπετε και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και η ψηφοφορία θα αρχίσει σε λίγα λεπτά μαζί με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.